Ευχαριστώ πολύ κύριε Βερζιά. Υποθέτω ότι και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε που είναι τόσο προσιλωμένε και αφοσιωμένε συμφωνούν. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν προ έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση και αν δεν διαφωνείτε θα διαβιβάσω στους αρμοδίους δικαιούχους και αποδέκτες τα όσα μόλις ψηφίσαμε.